Θα προχωρήσουμε τώρα στις ε, επεξηγήσεις ψήφου. Καλώ όλους τους βουλευτές ε, που θέλουν να φύγουν από την αίθουσα και που δεν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συζήτηση να φύγουν ησύχως. Σας ενημερώνω ότι έχω λάβει διάφορα αιτήματα για επεξηγήσεις ψήφου και μπορούμε να συνεχίσουμε όμως μόνο μέχρι τις 14.45 το αργότερο για να μπορέσουν οι υπηρεσίες να προετοιμάσουν την επανάληψη της συνεδρίασης στις 3. Όλες λοιπόν οι αιτήσει για αιτιολόγηση ψήφου θα, θα εξεταστούν ε, και οι υπόλοιπε θα υποβληθούν γραπτός όσες δεν μπορέσουν να γίνουν προφορικός. Ξεκινάμε την έκθεση Μόησα. Ησυχία παρακαλώ. Αναλαμβάνει στα γαλλικά ο Πρόεδρος. Όσοι δεν ενδιαφέρονται για τη συζήτηση παρακαλούνται να αποχωρήσουν. Πότσακ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένος ότι δεν θα γίνει ακουστή η φωνή μου, αλλά παρόλα αυτά θα μιλήσω. Χαίρομαι για την προσέγγιση που έχει επιτευχθεί με τη Μολδαβία. Από την εποχή που ήμουν ήδη μέλος της Επιτροπής Φιλίας Μολδαβίας-Πολωνίας αγωνιζόμουν για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε επιτύχει σήμερα είναι η κορονίδα της διαδικασίας προσέγγισης, όπως είπα και στη συζήτηση προηγουμένως. Mm. Η συμφωνία σύνδεσης με την Μολδαβία οδηγεί και σε μια φιλελευθερωποίηση σε ό,τι αφορά τις προξενικές ε, θεωρήσεις, το καθεστώς του παρτενέρ και επίσης προτιμησιακές ε, ρυθμίσεις για τα δασμολογικά θέματα επιτρέπει να δοθούν 50 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της Μολδαβίας. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορούμε να δώσουμε πολλά θετικά για τη Μολδαβία. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα και συγχαίρω και την ίδια τη Μολδαβία για τη μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ. Τσαμπάσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ υποστηρίζω τις προσπάθειες που έχουν γίνει για υπέρ της Μολδαβίας, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κέριο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Είναι απαραίτητο να υπάρξει λοιπόν μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Η Κομισιόν θεώρησε ότι δεν θα υπάρξουν θετικά αρνητικά αντιπολέσματα και από τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται, γιατί αυτό είναι και θέμα πολιτικής ευθύνης. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι πρόκειται για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Μολδαβία ελάχιστης ποσότητας που δεν θα επηρεάσουν καθόλου την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς της Μολδαβίας να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους και έτσι <clears throat> με τη χρηματοδότηση που δίνουμε η οποία είναι ασήμαντη. Θα βοηθήσουμε λοιπόν την, την δοκιμαζόμενη αυτή χώρα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με την ε, χειρονομία αυτή βοηθούμε και την αντιμετώπιση των βουλγαρικών μειονοτήτων στη Βουλγαρία και έτσι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε στη μοίρα της αυτή την ε, ε, μειονότητα. Ευχαριστώ. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Α, ζητώ συγγνώμη. Ε, κύριε Πρόεδρε, Είμαι και εγώ υπέρ αυτή τη αλλαγή ε, σε ό,τι αφορά τι αυτόνομε εμπορικέ ε, προτιμήσει για τη δημοκρατία τη Μολδαβία. Χαίρομαι που δίνουμε αυτή την υποστήριξη και στέλνουμε αυτό το σαφέ μήνυμα. Ότι η Μολδαβία δεν είναι μόνη τη, αφημένη στη μοίρα τη, δίπλα στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Μολδαβία θέλει να είναι εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα ε, ε, καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και απαντά με διάνοιξη των αγορών της για τα γεωργικά προϊόντα από τη Μολδαβία και τη βοηθάει για να μπορέσει να επιβιώσει οικονομικά και να μπορεί να έχει μια πολιτική ανεξάρτητη και στην εξωτερική πολιτική και ανεξάρτητη από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν είναι μόνο εμπορικό και οικονομικό το πλεονέκτημα αυτό, είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα Υποστηρίζουμε μια χώρα η οποία θέλει να έχει ε, ελεύθερη, περήφανη, ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Χαιρετίζω λοιπόν αυτό το βήμα και ελπίζω στο μέλλον η Μολδαβία να είναι ισχυρό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Κέλλη. Επίση έχετε το λόγο και στα κελτικά. Ε, στα αγωεδελικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ έλαβα μέρος σε αυτή τη συζήτηση χθε και ήταν μια πάρα πολύ θετική έκφραση υποστήριξη προ τη Μολδαβία αυτή η συζήτηση και χαιρετίζω την ηλυμένη απόφαση. Και πράγματι εγώ υπερψήφισα αυτή την απόφαση. 551 βουλευτές υποστήριξαν αυτή την απόφαση, μια μεγάλη πλειοψηφία και αυτό δίνει εμπιστοσύνη στο λαό της Μολδαβίας και ιδίως τους μικροπαραγωγούς οι οποίοι βασίζονται στην δυνατότητα εξαγωγής φρούτων Προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πια δεν έχουν δυνατότητες εξαγωγή προς την Ρωσία λόγω της πολιτικής του Πούτεν και των σμπύρων του. Χρειάζεται όμως να προχωρήσουμε και να δώσουμε νέες αγορές στους μικρούς παραγωγούς της Μολδαβίας. Και αυτό είναι ιστορική απόφαση. Και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό καταδεικνύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας όταν βρίσκονται στα δύσκολα. Είμαστε πολύ κοντά τώρα στα Χριστούγεννα και αυτό είναι ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δώρο. Ευχαριστώ πολύ. Ντεπρέ, ο κύριος Γιάρ έχει το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Έχω κάνει μια αίτηση και έχω πάρει την ε, απάντηση σε σχέση με την έκθεση αυτή που αναφέρουμε. Ναι. Αναφέρεται στην προηγούμενη έκθεση ο κ. Βουλευτή. Δεν είσαστε στον κατάλογο, αν θέλετε λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, οι βουλευτές από όλες τις παρατάξεις του Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι υπέρ των μέτρων που ενισχύουν την κυριαρχικότητα της ε, Μολδαβίας και την δυτικόστροφη αντιμετώπιση των Βεσαραβών. Υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις εδώ στην επέκταση της ενιαίας αγοράς σε αυτόν τον παρατιμιστέριο χώρο. Θα πρέπει να καταλάβουν όλη τη διαφορά μεταξύ της ε, ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελεύθερο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί τα συγχαίουν γιατί νομίζουν ότι δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε Ευρωπαϊκέ Αγορέ, αν δεν είσαστε τμήμα των πολιτικών δομών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μακεδονία, τα νησιά τη Μάχη, η Νορβηγία, η Ανδόρα, το ακριτικό Λιχτενστάιν είναι κομμάτια τη Ευρωπαϊκή Αγορά, αλλά είναι κομμάτια τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε νόημα η Μολδαβία να μην έχει απρόσκοπτο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Γιάρ, τώρα για την έκθεση Ντεπρέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα αξιοποιήσω την επεξήγηση μου για να επενέσω και πάλι την Επιτροπή Προπολογισμού. Διορθώσαμε ε, τον προπολογισμό για το 2014 και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις ε, για να αποφασίσουμε ένα προπολογισμό και για το 2015. Από τη μια όλα αυτά είναι απαραίτητα, από την άλλη είναι κάπως ενοχλητικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως χωλαίνει στη χρηματοδότηση μέσω των κρατικών συνεισφορών και με το ΦΠΑ που είναι ε, ήδη υπόρρη και από πρόστιμα, γι' αυτό χρειάζονται διορθώσεις. Αυτό που με ενοχλεί εμένα και με εξοργίζει ε, δεν είναι οι διορθώσεις που είναι απαραίτητες, αλλά αυτά που ζούμε κάθε χρόνο. Τα κράτη-μέλη κάθε χρόνο ξεχνούν να πληρώνουν εγκαίρως τις συνεισφορές τους και θα πρέπει κάθε φορά να τρέχουμε να ε, ε, προλαβαίνουμε ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο και για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 3. Κύριε Γιάρ, έχετε εγγραφεί και δεύτερη φορά η επεξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να συνεχίσω ακριβώς από εκεί που σταμάτησα. Θα ήθελα να παρακαλέσω απλούστατα γιατί με το προπολογισμό του 2014 και το διορθωτικό ε, του 2014 δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε όλοι και ενώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως τα κράτη-μέλη, όλοι τώρα να συγκεντρωθούμε σε αυτό, να δούμε τι θα γίνει με το backlog που είναι οι απλήρωτοι λογαριασμοί που συσσωρεύονται και δεν συσσωρεύονται επειδή δεν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να δαπανά χρήματα, ούτε σπαταλάει τα λεφτά. Απλούστατα τα κράτη-μέλη δεν καταβάλουν τις συνεισφορές τους. Ε, θα παρακαλούσα να εξοφληθούν αυτοί οι λογαριασμοί και να συμφωνήσουμε ε, για το τι μέλη γενέστε, να πληρώνουμε εγκαίρως τους λογαριασμούς και επίσης τα κράτη-μέλη εγκαίρως να καταβάλουν τις δικές τους συνεισφορές. Η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το επίπεδο των ε, μη πληρωμένων λογαριασμών, τα ΡΑΛ, αυξάνουν κάθε χρόνο. Έχουν φτάσει και έχουν ξεπεράσει τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ υψηλό αυτό το επίπεδο και ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ήδη σε μεγάλε δυσκολίε. Οποιασδήποτε ε, καθυστερήσει αυξάνουν την έλλειψη αξιοπιστία που νιώθουν πολλοί πολίτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό εγώ ενέκρινα τον τωρινό προπολογισμό, όπου προβλέπεται μια, ένα ποσό 4,2 δισεκατομμυρίων για να καλυφθούν οι ενεκρεμότητοι λογαριασμοί. Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας αυτό. για το τέταρτο διορθωτικό προϋπολογισμό. Η κυρία... Παγάσα Ορτουντούα ε, Ρουίθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τη Μεσόγειο έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να μιλάμε, αλλά δεν θα κουραστούμε μέχρι να είναι ικανοποιητική κατάσταση. 3.224 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο, ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σύμφωνα με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Αυτό είναι μία μόνο από τις πτυχές και τα πρόσωπα της περίπλοκης κατάστασης της μετανάστευσης στις χώρες μας. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις αιτίες, τις συνέπειες με σύνεση, με λογική. Αλλά να δούμε τις νόμιμες μεταναστευτικές ροές με βοήθεια προς τις χώρες καταγωγής και αντιμετώπιση της βίας ε, που ε, παράγεται από τη φτώχεια, τον ολοκληρωτισμό, τα αποτυχημένα και χρεοκοπημένα κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται απολύτω τη διαχείριση όλων αυτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μεταναστών. Να σκεφτόμαστε παγκόσμια αλλά να δρούμε τοπικά. Να είμαστε κοντά στην εκάστοτε τοπική πραγματικότητα, στην παραμεθόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ απόλυτα απαραίτητη μια καθολική και σφαιρική προσέγγιση μετανάστευσης. Ο κύριος Γιάρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε κλείσει τη διαδικασία του 2015 και δεν έχουμε το πρόβλημα της στενότητος ρευστότητος που φοβόμασταν και αυτό οφείλεται στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με τη σωστή επίτευξη συμβαστικών λύσεων εξασφάλισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις υποχρεώσεις τους. Έχουμε λοιπόν την ε, διαφορά αυτή ανάμεσα στις υποσχέσεις νέων προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως αντιμετωπίζουμε προβλήματα ρευστότητας και έχουμε πολλούς λογαριασμούς οι οποίοι παραμένουν από το παρελθόν. Και εδώ βλέπουμε όμως και ένα θετικό αποτέλεσμα πόσο καλός και αγαθός μπορεί να είναι ο κόσμος αν τα κάτι μέλη τηρούν τις υποσχέσεις τους και τις υποχρεώσεις τους. Βλέπουμε ότι έχουμε μειούμενο ε, ΑΕΠ έχουμε χαμηλότερα έσοδα από το, από το ΦΠΑ. Από την άλλη μεριά, τα πρόστιμα μα έχουν βοηθήσει να καλύψουμε αυτό το κενό. Πόσο πιο όμορφο και αγγελικό θα ήταν ο κόσμο αν τα κατημέλη πάντα συνεργαζόταν. Περνάμε στο πέμπτο διορθωτικό προπολογισμό. Ο κύριος Σόλτες έχει το λόγο. Δεν είναι παρόν. Ε, η κυρία Μπέγκιν. Δεν είναι παρούσα. Μωρέτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά τη συμφωνία για του προπολογισμού 2015 δεν θεωρούμε πως είναι επαρκές και εικονοποιητικός αλλά ως κοινοβούλιο που χρειάστηκε να το υπερψηφίσουμε λόγω της μεγάλης αίσθησης ευθύνη που μας διακρίνει. Η κυρία η σοσιαλίστρια κυρία Γουάρδια Ζαβάλ και επίση ο κύριος Ρέντζη μας είπαν ότι φτάνουν τα χρήματα. Όμως εμείς πιστεύουμε πω δεν φτάνουν γιατί το, το Συμβούλιο έχει πέσει θύμα ε, εθνικών εγωισμών Γερμανία, Γαλλία και ε, Βρετανία που θέλησαν να πνίξουν αυτή τη συμφωνία. Όμως το Κοινοβούλιο μπόρεσε να σταθεί στο ύψος του και να δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα πιο σημαντικά προγράμματα όπως ε, το Έρασμος και το Ορίζοντας 2020 όσον αφορά τις πληρωμές. Ωστόσο θα πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση ευφυής και λειτουργική όσον αφορά τη δημοσιονομική διαδικασία που διαρκώς δείχνει τα ωριά της. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα αυτό το διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2014 46,9 δισεκατομμύρια ευρώ κινητοποιήθηκαν για την επίγουσα βοήθεια προς την Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία για τις ε, θεομηνίες. Ε, ε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ζημίες και μόνο στην Κροατία οι πλημμύρες μας έχουν στοιχείς 291 εκατομμύρια σε ζημίες και ανάγκασαν πολύ κόσμο να εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Είναι πολύ λίγα τα κονδύλια που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε όλες τις ζημίες. Γι' αυτό χρειάζονται και άλλα ταμεία για να βοηθήσουμε τα θύματα. Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι θεομηνίες που έπληξαν πρόσφατα την Ευρώπη έπληξαν και τη Σλοβενία και την Κροατία και την Ελλάδα και προξένησαν τεράστιες ζημιές στις υποδομές. Επίσης, ε, αυτό αφορά τόσο ε, τις δημόσιες περιουσίες όσο και ιδιωτικές περιουσίες. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στις χώρες, γι' αυτό ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός να βοηθήσει για να αντιμετωπιστούν οι ζημίες. Στην Κροατία τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί θα είναι πολύτιμη βοήθεια ε, για τις περιφέρειές μας που επλήξαν περισσότερο. Thank you, Mr. Deputy Speaker. I Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη αντίδραση του νομοθέτη κανονικά σε μια κρίση είναι να πάει να πιάσει το πορτοφόλι του, αλλά κανονικά ε, βάζει το χέρι στο δικό σου πορτοφόλι. Δηλαδή, μόλις γίνονται τέτοιες ε, καταστροφές και θεομηνίες, ε, βάζουμε το χέρι στο πορτοφόλι των αλλωνών και έτσι δείχνουμε πάρα πολύ ευαίσθητοι και καλοί. Εάν σας συγκινούν όμως τόσο πολύ οι θεομηνίες και οι καταστροφές, βάλτε τα χέρια στις δικές σας τσέπες, στα δικά σας πορτοφόλια και δεν το λέω αυτό μόνο ηρωνικά και ρητορικά, αλλά μια από τις ε, ε, καταστροφές, διαρκώς πλημμύρες ε, συμβαίνουν στη Σλοβενία και στα Δυτικά Βαλκάνια γενικά. Ήδη το Μάιο είχε γίνει Σλαβωνία τέτοια πλημμύρα και καθάριζαν τις ζημιές με το φίλο Τόμασιτς που είναι τόσο πατριωτικός και κατά της διαφθοράς στην Κροατία. Καλύτερα να πα να βάλεις το χέρι σου, να πιάσει το φτιάρι, να κάνεις κάτι. Σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ καλύτερα παρά να βουτάς το πορτοφόλι των άλλων. Πρόεδρος, δεν μπορώ να επιτρέψω μπλε κάρτες, διότι δεν πρόκειται για συζήτηση. Πρόκειται μόνο για επεξηγήσει ψήφου. Περνάμε λοιπόν στην έκθεση Δεπρέ. το 7ο διορθωσχέδιο του δικού προπολογισμού. Κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Μετά από τις ε, πλημμύρες στη Βουλγαρία το 2014 πολλά χωριά έχουν καταστραφεί. Υπήρξαν δεκάδες θάνατοι. Έχουν καταστραφεί οι υποδομές επικοινωνίας και συγκοινωνίας και δεκάδες χιλιάδες άτομα χρειάστηκε να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους πρέπει εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουν όλα αυτά τα άτομα να επανέλθουν στη φυσιολογική του ζωή. Γι' αυτό εγώ <clears throat> ζήτησα από τις τοπικές αρχές να κάνω μια αξιολόγηση των ζημίων. <clears throat> από 13 περιφέρειες πήρα στοιχεία από διάφορους δήμους και όλα αυτά τα έχω διαβιβάσει στις εθνικές μας βουλγαρικές αρχές και η κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης θα μας βοηθήσει να ανοικοδομήσουμε τις υποδομές στην περιοχή μας όπου ζουν πάνω από 3,3 εκατομμύρια Βουλγάροι πολίτες, ο κ. Σαμπάφσκι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο... η έκθεση για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δοθεί μια οικονομική υποστήριξη στη Βουλγαρία πάνω από αυτήν η οποία παρέχεται αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ασήμαντη. Έχουμε πάνω από 300 εκατομμύρια ζημίες και παίρνουμε μονάχα 6 εκατομμύρια. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια υποστήριξη που να είναι ουσιαστικότερη και να αντιστοιχεί στη σημασία της αλληλεγγύης. Δεν μπορεί λοιπόν χώρες <clears throat> όπως η Βουλγαρία να παίρνουν έξι φορέ λιγότερη βοήθεια από μια γειτονική χώρα όπως η Σερβία η οποία δεν είναι μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρόλα αυτά παίρνει 60 εκατομμύρια υποστήριξη. Θα πρέπει λοιπόν να μην έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι με κατάφορο τρόπο θίγουν χώρε οι οποίε είναι φτωχότερε από του γειτονέ του. Νομίζετε ότι με 10 εκατομμύρια έχετε μπορέσει να καλύψετε ζημίες οι οποίες ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια. Η βορειοδυτική Βουλγαρία είναι το φτωχότερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο μηχανισμός αυτός δεν βοηθάει τις φτωχές χώρες, τις αφήνει να βγάλουν μόνες τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν είναι μηχανισμός λοιπόν αλληλεγγύης. Η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σημαντική και αυτή η απόφαση, 80 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για να βοηθηθούν η Κροατία, η Βουλγαρία και η Σερβία μετά τις μεγάλες πλημμύρες του Μαΐου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα κονδύλια αυτά για να ε, επαναρθωθούν οι ε, ζημίες που έγινε και να αποκατασταθεί η κατάσταση. Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε τη σημασία της πρόληψης και όχι της αποκατάστασης των ζημιών. Θα πρέπει να γίνουν έργα γιατί οι πλημμύρες είναι όλο και πιο συχνές στην Ευρώπη. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε ε, πόρους από τα επενδυτικά ταμεία και από άλλες πηγές για την πρόληψη έτσι ώστε στο μέλλον να μην έχουμε τέτοιου είδους θεομηνίες. Ο κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αυτό ο διορθωτικός προπολογισμό παριθμών 7 για το 2014 είναι υψής της σημασίας, διότι επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης και για την Κροατία, γιατί είχαμε τεράστιες ζημιές μετά από τις ε, πλημμύρες. Ε, εκατοντάδες χιλιάδες ε, σπίτια επλήγησαν και στην Κροατία και στους γείτονές μας, στην Βοσνία Ζεγοβίνη και στη Σερβία. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυσκολίες, τεράστια τα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν. 300 εκατομμύρια ευρώ ε, ε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς είναι οι ζημίες. Η Κροατία θα αντλήσει γύρω στα 9 εκατομμύρια για τις ομινίες και την κακοκαιρία και συνολικά 16 εκατομμύρια. Ε, νομίζω ότι τα χρήματα αυτά θα πιάσουν τόπο, θα ενισχύσουν και τις περιφέρειες που επλήγησαν ιδιαίτερα σφοδρά. Πίκουλα. Με ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σφοδρές αυτές οι θεομηνίες και για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης ακριβώς ε, ε, οι θεομηνίες ήταν εκείνες που μας ενέπνευσαν. Ε, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και είναι συμβολικό ο χαρακτήρας των ποσών που κατατίθεται. Ε, πρέπει να έχουμε πνεύμα αλληλεγγύη στην Ευρώπη, αλλά να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον αυτές τις καταστάσεις. Οι υποδομές μας είναι παλιές, ε, χρειάζονται ενίσχυση και μέχρι το 2020 η Κροατία θα πρέπει να επενδύσει 45 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κούνα, που είναι περίπου ε, ε, ο μισός προϋπολογισμός του κράτους. Μπορούμε να καταλάβουμε ε, τι δυνατότητες έχουμε. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης αλλά και άλλων ταμείων να βοηθήσουν τις χώρες ε, που ε, κινδυνεύουν. Τόμασιτς. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα φυσικά ε, αυτή την έκθεση και το διορθωτικό προπολογισμό και συμφωνώ με τους περισσότερους συναδέλφους της ομάδας μου ε, που μίλησαν για τους διορθωτικούς προπολογισμούς γενικότερα του 2014 και τον ε, προπολογισμό της Ένωσης για το 2015. Το ξέρω ότι ζητούμε περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία από τις χώρες μέλη που πρέπει να κάνουν θυσίες και να σταματήσουν αυτή την πρακτική να δαπανούν χρήματα που δεν έχουν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι ευρωβουλευτής από την Κροατία και γνωρίζω πάρα πολύ την κατάσταση επιτόπου. Είναι μια χώρα που έχει πληγεί πάρα πολύ από τις ε, πλημμύρες. Πολλοί συμπολίτε μας έχουν χάσει τα σπίτια τους. Οι συμπατριώτες μας ε, αντιμετωπίζουν ε, τεράστιες δυσκολίες και βρίσκουν τις συζητήσεις μας πάρα πολύ αφηρημένες χρειάζεται οπωσδήποτε βοήθεια. Και αυτό θα βοηθήσει και για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε στο νέο σχέδιο προπολογισμού 2015, ο κύριο Σόλτης. Λείπει. Μόντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον Οκτώβριο οι συνάδελφοί μου από το Labour και άλλοι ψήφισαν για να κάνει κάτι περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ένα παράδειγμα αυτό όμως όταν ο, η Φίλης έχει ε, ε, προσκομιτώθηκε σε ένα κομίτι. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει σημαντική πρόοδος εφέτος με την αντιστροφή πολλών από τις πιο καταστροφικές περικοπές του Συμβουλίου που θα είχαν θίξει μικρές επιχειρήσεις, μικρές κοινότητες και ερευνητικά κέντρα στην περιοχή μου. Δυστυχώ δεν είδαμε σωστή ανακατονομή των πόρων από την κοινή αγροτική πολιτική ή από τι μηνιαίε επισκέψει μα στο Στρασβούργο. Τι ωραίο μέρο, Αλλά αυτό δεν είναι η καλύτερη χρήση χρόνου και υλικών πόρων. Θέλουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια να χρησιμοποιούνται εκεί που υπάρχει πραγματική προσθέμενη αξία για του πολιτέ μα και σχέδια τα οποία ενισχύουν τον διεθνή ρόλο μα. Εγώ προσβλέπω στο να προχωρήσει ο προϋπολογισμός προς αυτή την κατεύθυνση το 2015. Δεν βλέπω τον κύριο Λούνες, την κυρία Γκίλ ούτε. Δίνω το λόγο στην κυρία Μωράτη. Ναι κύριε Πρόεδρε, παρά την έγκριση αυτού του προπολογισμού, πιστεύω ότι μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ας ε, θυμηθούμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι σοσιαλιστές και οι δημοκρατικοί, αλλά το Συμβούλιο ε, ακόμα μια φορά αποτέλεσε θύμα, έπεσε θύμα της ισχύω και της και, ε, επικυριαρχίας κάποιων χωρών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία. Ωστόσο καταφέραμε να επιτύχουμε κάτι σε σχέση με αυτές που είναι οι δεσμεύσεις που πρέπει να παραμένουν ε, ζωή για σημαντικά προγράμματα όπως το Έρασμος και το ορίζον 2020. Ωστόσο, παραμένει πάντα προτεραιότητα η δέσμευσή μας για μια ευφυή και λειτουργική μεταρρύθμιση του συνόλου της διαδικασίας μεταρρύθμισης ε, του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κινίτσι έχει τώρα το λόγο. Η κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρότι θεωρώ πως η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα, υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί η αύξηση των κορδιλίων σε σχέση με τον προηγούμενο προπολογισμό επιτρέπει να απευθυνθούν περισσότεροι πόροι, ακόμα και χαμηλό, αν είναι χαμηλότεροι από αυτούς που θα έπρεπε, σε κάποιες στρατηγικές ε, προτεραιότητες μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που έχει ε, ως στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η παρέμβαση υπέρ της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημαίνει ότι επενδύουμε στο μέλλον της Ένωσης και των πολιτών της, εντατικοποιώντας την καταπολέμηση της ανεργίας, της οποίας τα ποσοστά παραμένουν εξαιρετικά ψηλά, κυρίως για τους νέους, για ορισμένες περιφέρειες. Θεωρώ πως είναι θετική και η δέσμευση του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον διορθωτικό προπολογισμό του 2014, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνέχεια στις δράσεις της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα των θεομηνιών όπως αυτή που έπληξε τη Σαρδινή, για την οποία δόθηκαν 16 εκατομμύρια. Το λόγο έχει ο κύριος Πάλσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, της ομάδας του Γιόμπικ δεν μπορώ να πω ε, δεν μπορούσαμε παρά να καταψηφίσουμε τον προπολογισμό του 2015. Επαναλαμβάνεται η νέα νεοφιλελεύθερη, η ίδια νεοφιλελεύθερη στρατηγική και συνταγή του παρελθόντος. Ε, η πλειοψηφία κατέριψε, καταψήφισε όλες τις δικές μας τροπολογίες που ήθελαν να καταργήσουν αυτή τη νεοφιλελεύθερη πολιτική. 4,5% είναι η μείωση στον επταετή προϋπολογισμό και 8,4 στα ταμεία συνοχής. Τι σημαίνει αυτό. Οι λεγόμενες κεντρικές χώρες και οι περιφερειακές ε, βλέπουν το χάσμα το οποίο τις χωρίζει να διευρύνεται. Ωραία τα καλά λόγια που λέτε και επαναλαμβάνετε για την οικονομία, για την ανάκαμψη, για την Ενωμένη Ευρώπη. Οι αριθμοί όμως μιλάνε άλλη γλώσσα. Η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Συμφωνία για τον Προπολογισμό του 2015 επετεύθη κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής. Εγώ τον υποστήριξα γιατί ήταν σημαντικό στην αρχή του επομένου έτου, να έχουμε προπολογισμό και να μπορούν τα κράτη-μέλη να ε, καθησυχαστούν. Ο προπολογισμό του 2015 όμω δεν λύνει όλα μα τα προβλήματα. Περιμένουμε από τα θεσμικά όργανα να καταβάλουν μεγαλύτερε προσπάθειε για να ε, αντιμετωπίσουν αυτό το ξύτατο πρόβλημα. 142 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται στον προπολογισμό φέτο, αλλά αυτό σημαίνει σημαντική μείωση σε σχέση με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανερχόταν σε 146 δις. Ποιος θα πληρώσει τη διαφορά? Θα μεταφερθεί ένα τμήμα της το 2016. Πάντως θα πρέπει να εξοφληθούν οι απληρωτοί λογαριασμοί. Κύριος κορβέτ. Thank you. Year after year, some member states seem to pay far more attention πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία, λέει ο κύριο Κόρμπετ, ιδιαίτερη προσοχή στο επίπεδο των δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον προπολογισμό. Πολλοί χρησιμοποιούν αυτό για να γνωρίσουν το περιεχόμενο του προπολογισμού, αλλά τα δύο είναι Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο του προπολογισμού και όχι στο ύψο του. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για τα κονδύλια αυτά τη δαπάνη, όπου οι δαπάνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξοικονομούν χρήματα σε εθνικό επίπεδο, με τον αποφύγουμε τον διπλασιασμό των προσπαθειών και επιτυγχάνοντα οικονομία κλίμακο, θα φαίνεται πιο αποδεκτό και πιο χρήσιμο ο ευρωπαϊκό προπολογισμό σε όλου. Και γι' αυτό νομίζω το τμήμα τη έρευνα και ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προπολογισμού που είναι μια σαφής περίπτωση που μπορούμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τους πόρους μας για να έχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητάμε περισσότερο σε εσωτερικές εθνικές συζητήσεις και αυτό αφορά ιδιαίτερα και τη δική μου χώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Άρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Και εγώ υπερψήφισα το προϋπολογισμό του 2015 όπως και πολλοί άλλοι και εγώ θα προτιμούσε ένα μεγαλύτερο προπολογισμό, αλλά όλα αυτά είναι λεφτά φορολογουμένων. Καταψήφισε την τροπολογία 4, η οποία ζήτησε να διπλασιάσουμε ποσά με την, του προπολογισμού με την αύξηση τη συμβολή των χωρών που έχουν το μεγαλύτερο ΑΕΠ. Η Ιρλανδία είναι όμω μια χώρα η οποία έχει γονατίσει από το χρέο τη. Έχει το έκτο μεγαλύτερο χρέο στην Ευρώπη, το 28. Δεν μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε τι συνεισφορέ μα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επίση, καταψήφισα τροπολογία 5, γιατί ενώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Ήδη το κάνουμε αυτό μέσω τη πολιτική συνοχή και το Ορίζον 2020 κτλ. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα κάνουμε στον προπολογισμό μόνο με την υποστήριξη των διαφορετικών πόρων. Όπως είπαν πολλοί ομιλητέ, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα πάρουμε τα χρήματά μας, πόσο καλά και αποτελεσματικά τα κάνουμε όλα αυτά, αντί να ζητάμε συνέχεια περισσότερα, περισσότερα ε, χρήματα, σαν να ερχόμαστε από μυθιστόρημα του κυρίου Ντίκενς. Περνάμε για την πρόταση ψηφίσματος όσον αφορά τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. κυρία Φεράρα έχει το λόγο η ευρώπη έχει το καθήκον να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει στους πολίτες της ε, την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αυτό βέβαια ε, γνωρίζουμε τις προκλήσεις στην ασφάλεια στην οποία υπόκειται όλο ένα και περισσότερο η κοινωνία μας. Βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να καταδικάσουμε αυτή την αύξηση αυτού του φαινομένου που εξάλλου ε, εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ήπειρό μας. Ε, αναφέρομαι στι εγκληματικέ οργανώσει, των οποίων η πρώτη διέξοδο είναι οι χώρε οι οποίε πιστεύουν ότι είναι άνοσες. Θα πρέπει να γίνουν αρκετά και για την καταπολέμηση της μαφίας. Μία συνολική προσέγγιση πρέπει να έχουμε σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να ακολουθήσουν ε, οι πράξεις ε, πέρα από τις ανακοινώσεις. Θα πρέπει να προβούμε σε κάθε δυνατή νομοθετική ε, ε, διάταξη ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις εγκληματικές οργανώσεις τύπου μαφίας ε, αλλά και να προστατεύσουμε τους όσους δίνουν πληροφορίες για αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Γκίλ ούτε και δίνω το λόγο στην κυρία Κινίτσι. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα επαναλαμβάνει ότι η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν παράλληλα. Θα πρέπει να εγγυηθούμε το πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων, γιατί δεν έχει εξασφαλιστεί αυτό πάντοτε στο παρελθόν, να είναι αποτελεσματική όμω η ασφάλεια και φυσικά να ελέγχεται από τι διάφορε δικαιοδοσίε. Αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να είναι αποτελεσματική στρατηγική και με αυτό το στόχο και αναμένοντα την ανακοίνωση τη Κομισιόν για τη νέα στρατηγική εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ψήφισμα εντοπίζει κάποιες ε, προτεραιότητες στις οποίες συμμεριζόμαστε μεταξύ αυτών η ε, αναχέτηση του δουλεμπορίου, ε, οργανωμένο έγκλημα, ανακύκλωση βρώμικου χρήματος και ούτω καθεξής. Επίσης, συνεργασία ποινικού, των ποινικών δικαστηρίων ανάμεσα στα κράτη, χρήση μεγαλύτερη των διαφόρων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και ε, οι διάφορες εγγύσεις που θα πρέπει να δοθούν με βάση την οδηγία περί προστασίας των δεδομένων. Γι' αυτούς τους λόγους υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα. Δεν βλέπω τον κύριο Ντότζ μπορούμε να περάσουμε στο ψήφισμα για την ε, αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Φορέντσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως ε, πρόκειται για ε, μια μέρα πραγματικά σημαντική για το κοινοβούλιο μας. Ευχόμεθα να είναι μια στιγμή που θα σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή για την αντίσταση και για τον λαό της Παλαιστίνης, για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, για την ειρηνευτική διαδικασία, για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη και για τους δύο λαούς. 135 χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Εγώ καλώ όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες να ε, πάνε σε αυτές τα μέρη όπου θα μπορέσουν να διαπιστώσουν με τα μάτια τους την καταστροφή που έχει προκαλέσει ο πόλεμος ε, του, από το πλευράς του κράτους του Ισραήλ, ακόμα και τους περασμένους μόλις μήνες. Ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει διαφορετικό ρόλο εκεί ε, και ελπίζω πως αυτό το ψήφισμα θα είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω πραγματικά να είναι σημαντική αυτή τη στιγμή έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να μπορέσει πραγματικά να λειτουργήσει υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας των δύο λαών. Βαλίνα. Δεν είναι εδώ. Δεν υπάρχει, δεν είναι στην αίθουσα. Thank Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα γιατί είναι ένα βήμα προς αυτή κατεύθυνση. Ανεγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, του λαού και των συνόρων. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Η διεθνή ε, κοινότητα καθυστέρησε και είναι ένα θετικό βήμα προς την ειρήνη. Τα κράτη-μέλη όπως η Ιρλανδία θα πρέπει να ενωθούν και να ε, προστατεύσουν το χώρο της ε, του Παλαιστινιακού κράτου ε, με βάση τα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική ε, Ιερουσαλήμ. Ο Παλαιστινιακός ε, λαός έχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και αυτό εγγράφεται σε διεθνή ψηφίσματα επί 66 χρόνια. Το Sinn καλεί όλα τα μέρη να αποφύγουν οποιαδήποτε δράση που μπορεί να υποσκάψει την βιωσιμότητα και τις προοπτικές μιας δικρατικής λύσης. Θα πρέπει να σταματήσουν οι οικισμοί και να σταματήσουν οι επιθέσεις καθώς και οι καταστροφές της Παλαιστινιακής ιδιοκτησίας. Ευχαριστώ. Κάρθη. Υποστήριξα μαζί με τους συναδέλφους το ψήφισμα για το Παλαιστινιακό κράτος. Είναι ευπρόσδεκτο αυτό το βήμα αυτού του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο, η Ευρώπη, τα κράτη-μέλη χρειάζονται να κάνουν πολύ περισσότερα για να υποστηρίξουν τον Παλαιστινιακό λαό και να εξασφαλίσουν ότι το Παλαιστινιακό κράτος όχι απλώς αναγνωρίζεται, αλλά θα δημιουργηθεί, θα είναι ένα λειτουργικό και βιώσιμο κράτο. Είδαμε φέτο το καλοκαίρι τι έγινε με αυτή την άνευ προηγουμένου παράνομη ε, εξοργιστική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Ω εκλεγμένοι άρχοντες έχουμε ευθύνη απέναντι στους λαού τη Ευρώπη να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα ξανασυμβούν. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι ως ε, κοινότητα απέναντι στο Ισραήλ. Γιατί η άγνοια, η αδιαφορία τους για το διεθνές δίκαιο είναι άνευ προηγουμένου. Έχουμε κάνει ένα πολύ πολύ μικρό βήμα. Ε, πρέπει να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερα όμως. Σεμπαστιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι το δικό μας ψήφισμα, δεν είναι τέλειο ψήφισμα. Λείπει, για παράδειγμα, η σαφής καταδίκη των ε, συνεχώς παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από πλευράς Ισραήλ. Ωστόσο, υπερψηφίσαμε το ψήφισμα αυτή και μάλιστα με πάρα πολλές ελπίδες και με πολύ μεγάλη χαρά γιατί υπήρξε συνένεση. Αυτό μας χαροποιεί και παρά τις ατέλειες αυτό το ψήφισμα επιβεβαιώνει τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών λαών να υπάρξει κράτος της Παλαιστίνης. Το ψήφισμα αναγνωρίζει τα δικαιώματα και την ανάγκη του Παλαιστινιακού λαού, ο οποίος ζει έγκλειστος μέσα στα εδάφη του, να έχει δικαίωμα σε ένα κράτος αναγνωρισμένο από όλους για να μπορέσει ο Παλαιστινιακός λαός να προχωρήσει προς κοινωνική δικαιοσύνη και να έχει μέλλον. Το ψήφισμα καλεί την Ευρώπη να αναλάβει δράση, να είναι στην πρώτη γραμμή του διεθνού στερεώματο, να είναι παρούσα στην ειρηνευτική διαδικασία. Έχει έρθει πλέον η στιγμή να αναλάβουμε το ρόλο που μα αναλογεί. Ευχαριστώ. Σοϊντρόβα έχει το λόγο. Mm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο θα ήθελα να εξηγήσω γιατί δεν μπορώ να στηρίξω το ψήφισμα αυτό για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους θα ήταν βεβαίω επιθυμητή, κατά την άποψή μου, μόνο εάν είναι το προϊόν μιας συμφωνίας δύο μερών. Δηλαδή, εάν ήταν το, πρωινό, το προϊόν μιας κοινή συμφωνίας Ισραήλ και Παλαιστινίων, ο απότοκος της ειρηνευτική διαδικασίας. Το ψήφισμα που προτείνεται δεν είναι σαφές και θα μπορούσε να ερμηνευτεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό αποτελεί κίνδυνο, ειδικά στη σημερινή χρονική συγκυρία όπου ε, εκτιλήσεται η προεκλογική εκστρατεία στο Ισραήλ. Και γι' αυτό το λόγο δεν δίναμε να στηρίξω αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. La parola Δεν υπάρχει στην αίθουσα. Σκρίπεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναγνωριστεί το Παστινιακό κράτος. αλλά καταψήφισα το ψήφισμα για τους εξής λόγους, παρότι υποστηρίζω τη δικρατική λύση. Γιατί ε, θα παραβιάσαμε το 16-7 της συμφωνίας του 95 του Όσλο. Πρέπει να περιμένουμε ε, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Παρότι εμείς υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία ως μάρτυρας, ε, είναι σαν να αμφιβητούμε αυτή τη συμφωνία το 1995. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με την σημερινή κυβέρνηση μπορεί να θεωρηθεί ως ε, de facto αναγνώριση της, της τρομοκρατικής κυβέρνησης Χαμάς αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, σήμερα διάβασα κάτι στον τύπο που ανέφερε ότι για διαδικαστικούς λόγους η Ευρώπη αναγνωρίζει μια τρομοκρατική οργάνωση. Μετά από 13 χρόνια, έτσι, παρότι αναγνωρίζω το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού, η αναγνώριση του κράτους ε, σήμερα θα ήταν ένα επιπλέον άχθος για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η δήλωση μιλάει για την καταρχήν αναγνώριση, αλλά όλοι θα θεωρήσουν ότι πρόκειται για πλήρη αναγνώριση και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη νομίζω ότι και για τις δύο αυτές οντότητες θα ήταν αρνητικό, θα ήταν ένα βήμα προς τα πίσω. Σόλτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθ' όλη τη διάρκεια της, ιστορία, της ιστορίας της, έχει υποστηρίξει την ειρηνευτική λύση του Παλαιστινιακού προβλήματος και της σύγκρουση με το Ισραήλ. Και προσπαθήσαμε πάντα να βρούμε την καλύτερη λύση που θα θέσει τέρμα στην καθημερινή βία. Το κάνει επί δεκαετίε τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012 υιοθέτησε ένα ψήφισμα που έλεγε ότι ένας ειρηνικός διάλογος είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να διευκολύνει την μακροπρόθεσμη και οριστική επίλυση του προβλήματος και της σύγκρουσης. Σήμερα ακούσαμε τους λόγους για τους οποίους δεν θέλουν κάποιοι να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος. Ενώ η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα ήταν ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση και για την ειρήνη. Ε, ότι είναι ο μόνος τρόπος για να επιληθεί ειρηνικά αυτή, αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό υποστήριξα το ψήφισμα. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε με μεγάλη ε, πλειοψηφία ε, το ψήφισμα αναγνώρισης ε, του κράτους της Παλαιστίνης. Και χαίρομαι διότι γίνεται αναφορά και στη ψηφοφορία στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Επιτέλους το Κοινοβούλιο μας έχει μια κοινή θέση που σέβεται πολλές από τις ευαισθησίες και τα λεπτά ζητήματα όλου αυτού του προβλήματος. Ηγέτες από το ΕΛΚ, από τους σοσιαλιστές, από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, από τους πρασίνους, κατάφεραν να πετύχουν σε συμφωνία, σε ευρία βάση. Ναι, υπάρχουν διαφωνίες για, για την προθεσμία, αλλά είναι αυτό ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι συμβολικό και δείχνει πόσο υπέρ είμαστε της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους και της λύσης δύο κρατών επί τη βάση των συνόρων του 67. Είναι επίγον να λυθεί το υπάρχον πρόβλημα, να ανακοπεί η επέκταση των Ισραηλινών επικισμών. Οι Ισραηλινοί χρειάζονται ασφάλεια και οι Παλαιστίνοι χρειάζονται τα δικά τους σύνορα, το δικό τους κράτος. Ελπίζω ότι το ψήφισμά μας θα βάλει ένα λιθαράκι σε όλο αυτό το οικοδόμημα της ειρήνης. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Πίκουλα έχει το λόγο. Ε, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταρχήν αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, της ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης είναι μια ιστορική στιγμή, αλλά ένα βήμα μόνο δεν είναι η απόκτηση αυτού του καθεστώτος. Διάφορες ε, πολιτικές ομάδες εκφράστηκαν υπέρ της επίτευξης αυτού του στόχου όπου υπάρχουν διαφορετικές γραμμές αφετηρίας. Σήμερα γίνεται προσπάθεια να εξευρεθεί μια λύση για να μην υπάρξουν περαιτέρω βιοπραγίες. Και δεν βλέπω εδώ και την αναγνώριση της κρατικής οντότητας ως συνεισφορά περαιτέρω μαχών και σειράξεων, αλλά ως συνεισφορά για επίλυση του προβλήματος. Ως Ισραήλ δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς έναν ιδανικό εταίρο διαπραγματεύσεων. Όμως αναμένουμε από αυτό το ψήφισμα, με αυτό το ψήφισμα από τους Παλαιστίνιους να λάβουν υπόψη τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου και την λύση των δύο κρατών να προσπαθήσουν να την επιτύχουν με ειρηνική συνύπαρξη. Είμαι υπερήφανη σήμερα που υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση για να αποκτήσει κρατική οντότητα η Παλαιστίνη. Και πέρα από την, το ενδυναμωμένο κίνημα για την υποστήριξη του κράτους της ε, Παλαιστίνης, προσθέτουμε και τη φωνή μας από την Ιρλανδία με ένα ψήφισμα του Sinn Féin να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ε, από το Ισραήλ και να αναγνωριστεί η κρατική οντότητα της Παλαιστίνης. Όμως με την επιθετική επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη που έχουν σημαντικές επιπτώσεις εις βάρος των διαπραγματεύσεων είναι σημαντικό η διεθνή κοινότητα να υπογραμμίσει το ότι υποστηρίζει την κρατική οντότητα της Παλαιστίνης. Αυτό το ψήφισμα θα έστενε ένα ισχυρό μήνυμα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ειρηνική επίλυση του ζητήματος. Ευχαριστώ. Ζάνι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αυτό το ψήφισμα εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Όμως θεωρώ ότι εύθετο θα ήταν εκείνοι που απήχαν όπως εγώ να μπορέσουν να εκφράσουν την άποψή τους. Απήχα επειδή ήθελα να δείξω με τη στάση μου ότι έχω δισταγμούς να δεχθώ κάποια στοιχεία από αυτό το ψήφισμα. Κυρίως τις επιπτώσεις, τις συνέπειες αυτής της αναγνώρισης της κρατικής οντότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω η Ευρωπαϊκή Ένωση να, με πολύ μεγαλύτερο σθένος να αναλάβει δράση με τον ε, ρόλο που πρέπει να έχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ώστε να επιτευχθεί η λύση των δύο κρατών και μια μακρόβια ειρήνη που θα επιτευχθεί και πιστεύω ότι οι προσπάθειες ε, <clears throat> της ε, είπα της εκπροσώπου Μογαρίνη πρέπει να τύχουν της υποστήριξής μας. Αυτό θα απαιτήσει χρόνο φυσικά και συνεργασία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου των άλλων θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών φυσικά. Η αναγνώριση τώρα <clears throat> της ε, Παλαιστίνης με μονομερή τρόπο από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι θα οδηγούσε στο να υπαναχωρήσει, να οπισθοδρομήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Είναι ένα μέσο λοιπόν, ένα εργαλείο και όχι αυτός σκοπό η αναγνώριση αυτή. Ευχαριστώ. Με ακούτε? Καλώς. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην θεωρήσουμε, ας μην αναγνωρίσουμε με έναν τρόπο επονίδιστο. Πολλοί προσπάθησαν να παρεμποδίσουν αυτή την ψηφοφορία με ευρωσκεπτιστική ευρωσκεπτικιστικό και συντηρητικό τρόπο και καλό θα ήταν το Κοινοβούλιο να μην αφήσει την, να την ιστορία να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια του για άλλη μια φορά χωρίς να κάνει τίποτα. Και αυτό το αποφύγαμε. Ε, ξεκάθαρα είπαμε τι πιστεύουμε. Βεβαίω υπάρχουν κενά στο ψήφισμα, δεν γίνεται λόγο για του Ισραηλινού επικισμού, για τα εμπόδια στην ειρήνη. Ωστόσο, είναι ένα καλό ψήφισμα και ελπίζω το Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ε,

Ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα μάλλον θα διατάξει το πέρας των επικισμών μέχρι το 2016. Ελπίζω να είναι σε θέση να δώσει ένα τέλος σε όλα αυτά. Να είμαστε περήφανοι και εμείς και τα εθνικά κοινοβούλια που έχουν απαιτήσει την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα λοιπόν οι φίλοι μας ε, Παλαιστίνοι και Ισραηλινοί γνωρίζουν ότι με αυτό το περιστατικό, με αυτό το ψήφισμα είμαστε στο, πλευρό τους. Έχει έρθει η ελπίδα πλέον στην Ευρώπη και θα πρέπει να δοθεί η αναγνώριση στο κράτος της Πανελληνιστίνης, το οποίο ζητούν τόσο πολύ καιρό. Ο κύριος Γκίλ, ευχαριστώ πολύ. Το UKIP ε, είναι υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Προσωπικά πιστεύω ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα διευκολύνει τη διεθνή κοινότητα έτσι ώστε να λάβει σάρκα και οστά η λύση των δύο κρατών. Πιστεύω ότι μία, μία μέρα η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί. Ωστόσο, σήμερα ε, ψηφίσαμε ένα ψήφισμα το οποίο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει και εγώ δεν έχω καμία πίστη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε ε, τι κάνει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, στη Λιβύη και στην πρώην, στις χώρες της πρώην Ιουκοσλαβίας. Ο υπεριαλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια καταστρεπτική και αποσταθεροποιητική δύναμη στον κόσμο. Δεν μπορώ να τον ενθαρρύνω ούτε να τον στηρίξω και δεν πρόκειται και να το κάνω ε, το να αναγνωρίσει κανείς ένα κράτος ε, σημαίνει ότι ε, αναγνωρίζει την ύπαρξή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητα να αναγνωρίσει κράτη όπως έγινε στην περίπτωση του Σομάλιλαντ. Επομένως δεν μπορούμε να ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά ε, με, σαν να ήταν κράτος γιατί δεν είναι. Μόνο κράτη έχουν την αρμοδιότητα να αναγνωρίσουν κράτη. Τζενόφσκι έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που προσπαθήσατε να διατυπώσετε σωστά το όνομά μου. Ευχαριστώ. Αυτό το ψήφισμα που δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω, διότι αυτό το κείμενο δεν μπορεί να επιλύσει κανένα πρόβλημα. Το σημερινό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου έχει ελλείψεις και δεν είναι σωστό. Ήδη προηγούμενα το είχα αναφέρει και πρέπει να το πω ότι εδώ όλο αντισημιτικές δηλώσεις ακούγονται και δηλώσεις κατά του Ισραήλ. Γι' αυτό αυτό το ψήφισμα θεωρώ ότι δεν συνεισφέρει υπέρ της ε, ειρηνευτικής λύσης ε, μεταξύ Πανιστινίων και Ισραηλινών. Mijn ε, partij N-VA heeft deze resolutie gesteund. Το κόμμα μου αυτό το ψήφισμα το υποστήριξε και αυτό για δύο λόγους. Όταν γίνεται συζήτηση για την Παλαιστίνη ως ε, κρατική οντότητα, είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς μαύρο-άσπρο μεταξύ δύο άκρων δηλαδή. Πρόκειται για την ασφάλεια και επιτέλους πρόκειται και για τον εκδημοκρατισμό και την δημοκρατία την ίδια, ίδια για την αυτοδιάθεση των λαών. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την δυνατότητα αυτή των Παλαιστινίων για μια λύση δύο κρατών όταν παράλληλα βαίνει εκ παραλλήλου με την διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και με την υποστήριξη και κάλυψη μέσω της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών εταίρων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν, πώς η συγκυρία θα μεταβληθεί και θα εξελιχθεί, πώς θα υπάρξει μια κυβέρνηση με αρμοδιότητες από πλευράς των Παλαιστινίων επί του συνόλου της επικράτειας ε, του Παλαιστίνης με τα σύνορα του 1967. Μόνο έτσι μπορεί να είναι μακροβια ειρήνη. Φέτη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα εγώ διότι αντανακλά πιστεύω και την δική μου άποψη και την άποψη των μελών του ΕΛΚΑ. Είμαστε υπέρ μιας λύσης ε, των δύο κρατών με ειρηνευτικές, με ειρηνικές διαδικασίες. Απαιτείται σωστή λειτουργία και δίκαια λειτουργία και η απόρριψη και καταδίκη ε, τρομοκρατικών οργανώσεων καθώς επίσης ε, και των φονταμενταλιστών. Η υποστήριξη τώρα από πλευράς της Χαμάσα ε, εμποδίζει μια λύση καθώς επίσης και οι επιθέσεις εις βάρος του Ισραήλ και η χρήση του ιδίου του λαού των Παλαιστινίων δηλαδή από την Χαμάσα βλάπτει τους Παλαιστίνιους και παρακολεί τη διαδικασία. Πρέπει η ειρήνη να είναι προϋπόθεση για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών. Ταυτόχρονα όμως και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις με βάση την, ε, τα όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση της Γενέβης ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα ήθελα να ζητήσω οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, να συνεχιστούν. Να θα διασφάλιζε αυτό και την ασφάλεια του Ισραήλ και της των Παλαιστίνιων και θα διασφάλιζε επίσης και μια δυνατότητα ειρήνης στην επικράτηση επικράτεια αυτή. Ο Ζάχραντι παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για τα θέματα αυτά και για την Παλαιστίνη έγινε ένα λάθος πρέπει να πω και αυτό για δύο λόγους. Εκ νέου το Ευρωκοινοβούλιο αναμίχθηκε σε θέματα και αρμοδιότητες που δεν το αφορούν και δεν έχει αρμοδιότητες. Δεν έχει αρμοδιότητες και εξουσίες η Ευρωβουλή και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναγνώριση μεμονωμένων κρατών. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα αυτό, πρέπει να παραδεχθούμε. Τα επιμέρους κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι διαφορετικά μεταξύ τους και προσπαθεί εδώ το Ευρωκοινοβούλιο σε μια συνολική λύση ισοπεδωτικά να αντιμετωπίσει τα πράγματα με ίδια μέτρα και σταθμά. Δεν γίνεται αυτό. Εξάλλου φοβούμε ότι τα ακραία στοιχεία από πλευρά των Παλαιστινίων θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν με ένα τέτοιο ψήφισμα από πλευρά μα. Διότι η Χαμά, για παράδειγμα, σε σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση και τον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, θα μπορούσε να θεωρηθεί με την αφαίρεσή τη από αυτόν τον κατάλογο ω υποστήριξη των Παλαιστινίων. Και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτού που χρησιμοποιούν τη βία. Γι' αυτό αυτό ήταν λάθο σήμερα. Johnson. Στηρίζω τη λύση δύο κρατών, όπως και το κόμμα μου. Ωστόσο, πώς μπορούμε να ψηφίσουμε αναγνωρίζοντας το κράτος μιας χώρας, της Παλαιστίνης, όταν ε, έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση παραδεχθεί ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα να το κάνουμε. Θα πρέπει να σταματήσει η ζημιά που γίνεται στη χώρα μου και επεκτείνετε τη ζημιά πέρα από τα σύνορά σας, ενώ δεν έχετε καθόλου τέτοιο δικαίωμα να το κάνετε. Ε, ε, Σέιμουρ, δεν θα απολογηθώ επειδή επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, εγώ και ο Τζίμιου Συνάδελφο, συνάδελφος ε, ε, θέσαμε θέμα διαδικαστικό. Ένα email μιας αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δήλωση ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει το κράτος, αλλά σήμερα αποδεικνύεται το αντίθετο. Δεν ξέρει η δεξιά τι πει η αριστερά. Δηλαδή, ό,τι και να γράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά στερείται νοήματος και ουσίας. Αυτή είναι η αποψή μου. Ευχαριστώ. James. James, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι ένα θέμα που πραγματικά δημιουργεί πολλές συγκινήσεις και αυτό συνέβη ε, σήμερα εδώ. Οι προθέσεις ήταν σίγουρα πολύ καλές, όμως η διαδικασία ήταν ελληματική, εξού και απήχα. Δεν μπορώ να στηρίξω μια πρόταση ψηφίσματος ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμφωνήσει επί της αρμοδιότητάς της και άρα δεν έχει την, το κύρος, ε, επισήμως δεν δύναται να κάνει κάτι τέτοιο τελικά υπονομεύονται οι προσπάθειες να λυθεί η σύγκρουση και θα μπορούσε ε, να ε, ε, ενταθούν και να οξυνθούν οι συγκρούσεις. Δεν μπορώ να αποδεχθώ το συμβολισμό υποτίθεται και τις εκ των υστέρων υπέρ της επίλυσης του προβλήματος. Δεν βοηθάει αυτό τους Παλαιστινίους. Η αποχή λοιπόν με αυτά τα κριτήρια είναι ο δρόμος που διάλεξα και το συνεχίζω να το υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Coburn. Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα το ψήφισμα αυτό αναγνωρίζοντας ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 3 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγραψε στο Τζιμ Καρέι τον συνάδελφό μου από το UKIP, και εξήγησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναγνωρίσει το Σομάλιλαντ ή οποιοδήποτε άλλο κράτος και ότι αυτό είναι προνόμιο των εθνικών κρατών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μπορούν να αναγνωρίσουν κράτη. Επομένως η αναγνώριση υποτιθέμενη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης του κράτους της Παλαιστίνης είναι παράνομη και οτι αυτο ειναι προνομιο των εθνικων κρατων της ευρωπαικης ενωσης τα κρατη μπορουν να αναγνωρισουν κρατη επομενω η αναγνωριση υποτιθεμενη απο πλευρας ευρωπαικης ενωσης του κρατους της παλαιστινης ειναι παρανομη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει παραδεχθεί γραπτός και εσείς θα έπρεπε να το είχατε καταψηφίσει αλλά δεν το κάνατε. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα πρέπει να γίνεται ή οποιοδήποτε άλλο κράτος από τα κράτη τα ίδια αυτά και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι έχουμε υπερβεί τα εσκαμένα, Ίσως ένας ε, πιλότος ο οποίος πραγματικά έχει συνέστηση του πώς οδηγεί και πώς πιλοτάρει το αεροπλάνο θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάντως σίγουρα όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο καλά θα κάνει να ασχοληθεί με τα ελλείμματα, με την Ευρώπη που καταραίει και όχι με θέματα τα οποία είναι τελείως εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτως του. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ διάβασα το κείμενο και να μην μιλάτε εσείς για την αρμοδιότητά μου. Εγώ διάβασα τι αρμοδιότητέ μου. Διάβασα το κείμενο του ψηφίσματος, έτσι, και ήταν πολύ σαφέ. Δεν υπάρχει καμία αναγνώριση ουσιαστική. Είναι μια υποστήριξη υπέρ τη διαδικασία αναγνώριση. Είναι ένα πολιτικό κείμενο και δεν έχει καμία νομοθετική εξουσία. Εγώ σα παρακαλώ απαντάω τώρα. Σα παρακαλώ. Περνάμε στον επόμενο μιλητή. εκτό μικροφώνου η απάντηση. προχωρούμε τη συζήτηση και πάμε στο χάλιβα. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Καστάντος σας Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά 67 χρόνια οδυνών, θανάτου και προβλημάτων, μία από τις πιο μακρές ε, και σκοτεινές σελίδες ιστορίας είναι ακόμα ζωντανή στη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε ότι αυτό το ψήφισμα σε καμία περίπτωση δεν είναι ε, η κορονίδα στην ενευτική διαδικασία που όλοι θέλουμε. Αλλά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και χαίρομαι για την ευρεία πλειοψηφία που εξέφρασε αυτό το κοινοβούλιο υπέρ του ψηφίσματος. Είπαμε ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην αναγνώριση, την οποία κάνουν τα κράτη-μέλη βέβαια, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει με αρμονικό τρόπο, όχι, όχι κακόφωνα, να αναγνωρίσουν αυτό το κράτος. Και αυτό ε, θα είναι δουλειά ε, που θα κάνει βέβαια, θα πρέπει να παίξει και η ύπατη εκπρόσωπος το δικό τη ρόλο. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ένα Παλαιστινιακό κράτο, ούτω ώστε να υπάρξει ασφάλεια και για τα δύο κράτη. Να είναι ένα κράτο δικαίου και να συμφιλειωθούν οι διάφορε φράξει, να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή η αναγνώριση θα είναι ε, δύσκολη. Τα λεφτά δεν φτάνουν. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε να επικρατήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη οι εξτρεμιστές. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ε, τα επόμενα χρόνια και ας μην γελιόμαστε. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος για το Χάλιβα. Φορέντσα. Με μικρόφωνο κατά προτίμηση. Είναι ανοιχτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα του Χάλιβα, όπως ξέρετε, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για μας. Και λόγω των πρόσφατων προβλημάτων της συντηρουργίας της Ιταλίας. Στον Τάρανδο, ε, στο Πιουμίνο και σε άλλες πόλεις. Εμείς συνεισφέραμε στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο και παρουσιάσαμε και μια προφορική ερώτηση μετά από την υπόθεση που συνέβη στο Τέρνη στην Ιταλία. Συζητώντα με τι τις των εργαζομένων που ήρθαν στις Βρυξέλλες και συνεχεία στο Στρασβούργο. Συνεργαστήκαμε και δουλέψαμε για να βελτιώσαμε το κοινό κείμενο. Τελικά όμως δεν μπορούσαμε να το υπερψηφίσουμε γιατί νομίζαμε ότι βάζει το θέμα του Χάλιβα στο investment package, στο πακέτο επενδύσεων του Juncker και μέσα σε μια ε, ιδεολογία ανταγωνιστικότητας που δεν μας πείθει. Εμείς θεωρούμε ότι Πρέπει να διατηρήσουμε το χάλιβα ως στρατηγικό στοιχείο στην παραγωγική διαδικασία της Ευρώπης. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όμως το κοινωνικό dumping και το περιβαλλοντικό dumping και να γίνουν σοβαρές οικολογικές μετατροπές, ούτως ώστε οι εγκαταστάσεις όπως του, τάραν, του ταράνδου που προκαλεί και θανάτους αλλά και καρκίνους να σταματήσουν να λειτουργούν. Εγώ είμαι από το Μίλτσμπορο ε, που υπάρχουν χαλιβουργίες ε, και όπου έχουμε ε, βιομηχανίες εντάσσεως εργασίας και χαλιβουργικές. Το 2009, το 2010 η κοινότητά μου αγωνίστηκε για να σώσει τη χαλιβουργία μας. Δεν θέλαμε απλώς να κρατήσουμε την βιομηχανική υποδομή μας. Χρειαζόμαστε επενδύσεις ε, σε, και στην υποδομή αλλά και σε εγκαταστάσεις που βελτιώνουν το περιβάλλον. Ε, και χρειαζόμαστε ε, χάλιβα που να μην περιέχει πολύ άνθρακα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης βιομηχανικές μονάδες για τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. εκεί, αν δημιουργηθούν, θα, αυτοί, αυτές οι εγκαταστάσεις θα φτιαχτούν 4.000 ε, θέσεις απασχόλησης και θα υποστηριχθούν άλλες 24.000. Με αυτόν τον τρόπο και το εργατικό δυναμικό και η βιομηχανία θα, θα εμπλακούν και καλό είναι να εφαρμόσουμε και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τζουφρίντα, θα ήθελα να σας πω ότι οι δηλώσεις ψήφου για τη Μεσόγειο θα γίνουν αύριο, μετά την ψηφοφορία. Γιατί στις 12.45 θα πρέπει να σταματήσω την ε, Ολομέλεια, ούτω ώστε να προετοιμάσουμε την επόμενη Ολομέλεια που θα ξεκινήσει ακριβώς στις 3. Τζουφρίντα. Η κυρία Τζουφρίντα. Ευχαριστώ. Ο τομέας του χάλιβα στην Ευρώπη έχει έναν ουσιαστικό ρόλο και είναι ζωτική σημασία για πολλά κράτη-μέλη. Και είναι λογικό που είναι προτεραιότητα τη βιομηχανική πολιτική Λόγω της διάστασης και λόγω της σημασίας για την απασχόληση τον καθιστούν σημαντικό και για την κοινωνική πολιτική. Η ισορρογική βιομηχανία μπορεί να δημιουργήσει 350, έχει μάλλον 350.000 θέσεις απασχόλησης άμεσες. Ε, Επομένω, πρέπει να μιλήσουμε για αγορέ, για ζήτηση, για ανταγωνιστικότητα, για εισαγωγέ και για εξαγωγέ. Είναι ακόμα όμω πιο σημαντικό και ίσω προτεραιότητα να μιλήσουμε για την προστασία και την κοινωνική ευθύνη όλα αυτά που λειτουργούν για τη βιομηχανία για να ανανεωθεί σε μια στιγμή κρίσης δεν πρέπει να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Ε, καταστροφές, ε, επανεγκαταστάσεις δεν μπορούν να βαραίνουν τους ε, εργαζόμενους. Το καθήκον μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν όταν ασχολείται με τη βιομηχανία να μην ξεχνά ποτέ τον κοινωνικό διάλογο. Όταν αυτά ευχαριστώ. Όταν αυτά που έκανα ως Επίτροπος ε, ασχολήθηκα με το θέμα του Χάλιβα και οτιδήποτε έκανα το έκανα και με τη συνεισφορά των συνδικάτων. Κάπερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά τα τελευταία έτη στην Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία χάπολε στι 40.000 θέσει απασχόληση. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω χιλιάδε θέσει απασχόληση που θα απολευθούν ακούγοντα τον πρόεδρο των Χαλιβουργών σε μια συνέντευξη στα όσα είπε. Πρόεδρε, η μεγαλύτερη χαλιβουργία στην πίνακη και είχε και αντίκτυπο στο αμέσα αυτό διότι ε, θα μετεγκατασταθεί στις ΗΠΑ λέει. Ανέφερε λόγους για την μετεγκατάσταση, την υψηλή φορολογία στην Αυστρία, υψηλά ενεργειακά κόστη, καθώς επίσης και έλλειψη πολιτικής βούλησης για μεταρρυθμίσεις από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστρίας. Είναι επίσης ε, πολύ δαπανηρές ε, οι ε, προδιαγραφές, αυστηρές προδιαγραφές για την έκκληση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και για την αγορά πιστοποιητικών ε, ε, ρήπανση τη εμπορία τρύπων. Όλα αυτά επιβαρύνουν την βιομηχανία στην Ευρώπη και οδηγούν στην αποβιομηχανοποίηση τη Ευρώπη. Οι Αμερικανοί το αντίθετο, η Αμερικανική κυβέρνηση επαναζωογονούν την δική τους βιομηχανία. Στην Ευρώπη δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια συμφωνία επ' αυτού λοιπόν από πλευράς Ευρώπης. Γι' αυτό υποστηρίζω την πρωτοβουλία του ψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία και το πρόγραμμα δράσης Τη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να επαναζωογονηθεί στην βιομηχανία τη Ευχαριστώ. Ανατού, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά ε, είμαστε ενώπιον των καλών προθέσεων της γραφειοκρατίας της Βρυξέλλες. Η χαλιβουργία στη Γαλλία έχει πληγεί, τα εργοστάσια συνεχώς κλείνουν και οι λίγες επιχειρήσεις που επιβιώνουν εξαγοράζονται από Ινδικές ή Κινέζικες πολυεθνικές. Στη Γαλλία η παραγωγή σε 30 χρόνια έχει πέσει κατά 40% ενώ η ζήτηση αυξανόταν. Αυτό είναι άμεση συνέπεια της πολιτικής των Βρυξελών, μια πολιτική η οποία ακολουθείται εδώ και δεκαετίες κατάργηση των ε, τελωνιακών εμποδίων, ε, ελεύθερο εμπόριο χωρίς καμία, ε, κανένα όριο. Και τελικά ό,τι προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά να καλύψει κάποια κενά ενώ το, και κάποιες τρύπε ενώ το καράβι συνεχώς βάζει νερά είναι εμπεγμός των υπαλλήλων των εργαζομένων. Θα πρέπει οι θύνοντες να ασκούν πολιτική η οποία να εξυπηρετεί τους λαούς και όχι το κεφάλαιο και τα χρηματιστήρια. Ευχαριστώ. Γκασπάρα, δεν νομίζω ότι είναι εδώ. Μπίλντε, ούτε. Γκρίφιν. Όποια, όλη η οικονομική ανάκαμψη εξαρτάται από μια ισχυρή κατασκευαστική βιομηχανία και η ευρωπαϊκή χαλιβουργία θα πρέπει να είναι μια βιώσιμη και επικερδής βιομηχανία. Συνυπέγραψα αυτό το ψήφισμα γιατί αυτά που κάνει η Κομισιόν για να προωθήσει τη βασική βιομηχανική παραγωγή σε όλα τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσει τις θέσεις απασχόλησης είναι πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν πρέπει να προωθήσει και να προστατεύσει ε, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ε, και περιβαλλοντικά πρότυπα σε όλη την Ευρώπη και να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα πρέπει να μην ξεχνά την ε, κατεπίγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί μια βιώσιμη ε, οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρωκα ε, και να χρησιμοποιήσει και την τεχνολογία δέσμευση και αποθήκευσης του άνθρακα. Γι' αυτό καλώ την Κομισιόν να δεσμευτεί να αναπτύξει υψηλής ποιότητα ενεργειακά αποδοτικά και κοινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες, να προωθήσει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις απασχόλησης στα πλαίσια της βιομηχανικής πολιτικής. Θα λάβει τον λόγο η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε υπέρ του ψηφίσματος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς επειδή θεωρούμε ότι η σοβαρή κατάσταση της χαλιβουργίας στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα του να, πωλείται, να ε, ξεπουλιέται αυτή η βιομηχανία και όχι να υπάρχει πραγματική ανταγωνιστικότητα. Στην Ισπανία οι ε, επιχειρήσεις υψηλής πρόσθετης ε, αξίας αντιμετωπίζουν απειλές κατάσταση από μεγάλες ομάδες υπερεθνικών, πολυεθνικών εταιριών. Αυτό πραγματικά οδηγεί σε πάρα πολύ σκληρές προσαρμογές. Από την άλλη πλευρά παραμένει αδρανής η Ευρώπη όσον αφορά τις μεγάλες καταχρήσεις των ολιγοπολίων. Από την άλλη πλευρά έχουμε επίσης ε, και ε, τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών θεωρούμε ότι η απάντηση στην βιομηχανική κρίση περνά μεταξύ άλλων με την ανάκτηση της δημόσιας ε, διαχείρισης όσον αφορά αυτούς τους στρατηγικούς τομείς με προγράμματα επενδύσεων ε, και επιχορηγήσεις ώστε να μπορέσουν αυτοί οι τομείς να είναι δυναμικοί και αποτελεσματικοί από το, την Ευρωβουλή εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τους εργαζόμενους ε, της Αλκόα, της Group και που δίνουν μάχη και αγώνα αυτή τη στιγμή για την απασχόληση και την εργασία τους και την ίδια τη βιομηχανία τους. Ευχαριστώ. Κινίτσι παρακαλώ. Κινίτσι. Ευχαριστώ. Ο τομέας του Χάλβα ήταν για την Ευρώπη πάντα ε, ένας από τους βασικούς ε, στρατηγικούς οικονομικούς τομείς. Και είναι αναμφίβολο ο κεντρικός ρόλος που αυτός ο τομέας έπαιξε στο παρελθόν και που έχει ακόμα για την ανάπτυξη και την ε, οικονομική ανάκαμψη. Όμω αντιμετωπίζει σοβαρέ δυσκολίε σχεδόν σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το ψήφισμα που μόλι ψηφίσαμε, ζητάμε από την Κομισιόν να εκπονήσει μέτρα και να προσαρμόσει τι πολιτικέ για να επανεκκινηθεί ο κλάδο, να γίνει ανταγωνιστικό και να αποφύγουμε λόγω τη παρατεταμένη κρίση να οδηγήσουμε σε μετεγκα... οδηγηθούμε σε μετεγκαταστάσεις των επιχειρήσεων του κλάδου. Ζητάμε ένα ειδικό λοιπόν σχέδιο ή πρόγραμμα για το Χάλιβα, ε, που θα εξασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος και ένα πακέτο οικονομικών ε, εργαλείων που θα επιτρέψει ε, στον κλάδο να ξαναπαίξει σημαντικό ρόλο και να είναι ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν υπερψήφισα το κείμενο. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση, η κυρία Σπυράκη. Okay κύριε πρόεδρε υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος την οποία και συνυπογράφω γιατί θέλω να υποστηρίξω τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο χάλιβας στην ευρώπη στην ελλάδα στην ελευσίνα στη μαγνησία στη θεσσαλονίκη. με βάση τα επίσημα στοιχεία της ένωσης χαλιβουργιών ελλάδος η συνολική παραγωγή το 2012 έπεσε σε σχέση με το 2007 κατά. 58%. σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση δηλαδή το δύο η εγχώρια ζήτηση έπεσε 82%. έχει δηλαδή επιστρέψει στα επίπεδα του 1962 ενώ οι ελληνικές εξαγωγές στο χάλιβα έχουν μειωθεί κατά 59% μόνο την περίοδο 2011-2014. Θέλω να σας πω ότι την ίδια ώρα οι τραπεζικές υποχρεώσεις για τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες χάλιβα στην Ελλάδα ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι δραματική πρώτα απ' όλα για τους εργαζόμενους εκεί. κατά συνέπεια νομίζω πως είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους ώστε να μειωθεί και η απόσταση ανάμεσα στο κόστος στο ενεργειακό κόστος στα κράτη μέλη και επίσης να φροντίσουμε ώστε να δημιουργηθεί και να προωθηθεί άμεσα ένα εμπορικό σχήμα ένα εμπορικό σήμα για δίκαια προϊόντα χαλιβουργίας κατασκευασμένα στην ευρώπη. ευχαριστώ. Σταματούμε μέχρι τις 3 η ώρα.